Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα όλους σας, ε, περίπου όλους σας, δεν είσαστε όλοι εδώ, να σας καλωσορίσω. Ορισμένα από εμάς είναι ήδη στην ώρα τους. Ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό κανόνα για το μέλλον. Αν κάποιος από εσά θέλει να λάβει το λόγο, μπορούμε να σας γράφουμε στον κατάλογο των ομιλητών και έτσι θα έχετε την ευκαιρία πρώτη να λάβετε το λόγο, ο έχετε τελευταίος παίρνει το λόγο μονάχα τελευταίος. Ο κύριος Γκίρεκ. Έτσι θα υπάρχει και ένομο συμφέρον να ερχόμαστε νωρίτερα. Θέλω λοιπόν να χαιρετήσω ιδιαίτερα την ε, κυρία Γκίγκαν Κουίν, την αρμόδια επίτροπη που για τα θέματα έρευνας, η οποία είναι ακριβώς στην ώρα της και έρχεται στην κατάλληλη στιγμή να μας πληροφορήσει για τα θέματα της αρμοδιότητάς της. Χαιρόμαστε επίσης για το γεγονός ότι υπάρχει ένα, θα μας πείτε και για ένα σχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο στα, στον τύπο, στα μέσα ενημέρωσης. Χαιρόμαστε λοιπόν πολύ για την παρουσία σας και σας δίνουμε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες καθώς και κύριοι, την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανίας, αναρωτιόμουν πώς θα ήταν να κάθομαι δίπλα σας. Φαίνεται ότι είναι πολύ ευχάριστο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία αυτή να ανταλλάξουμε απόψεις για το πρόγραμμα εργασίας για την Κομισιόν στον τομέα της έρευνας, της και της επιστήμης. Το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2010 στον τομέα της επιστήμης, κοινοτομίας και έρευνας θεσπίζει σημαντικές πρωτοβουλίες για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020 για ευφυά και βιώσιμη ανάπτυξη. Το σχέδιο αυτό καινοτομία θα θεσπίσει του τρόπου με του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την διακυβέρνηση σε επίπεδο Ευρω... και τι κυβερνήσει ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθήσουν τα θέματα καινοτομία και έρευνα για την ατζέντα του 2020, ώστε να δημιουργηθεί μια ένωση καινοτομία. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα μέλη τη Επιτροπή σα. Εγώ έχω αναλάβει το χαρτοφυλάκιο αυτό από τα χέρια του Μανουέλ Μπαρόζο για να προωθήσω αυτό το σχέδιο καινοτομία και είμαι επικεφαλή μια ομάδα Ευρωπαίων Επιτρόπων που τα χαρτοφυλάκια του άπτονται τη έρευνα και τη καινοτομία. Επίση, κάνω διαβουλεύσει με όλου του εμπλεκόμενου στα θέματα τη καινοτομία, στην έρευνα, στην αγορά κτλ. για να δούμε ποιε συγκεκριμένε δράσει θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτό το σχέδιο. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιε είναι οι απόψει όλων των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλων των μελών της Επιτροπής Βιομηχανίας για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε με το σχέδιο αυτό. Χρειαζόμαστε να άρουμε όλα τα εμπόδια για την επίτευξη μιας κοινή αγοράς καινοτομία. Επίσης, θα παρουσιάσει, ο κύριος, θα παρουσιάσει ο κύριος Μπαρός το σχέδιο αυτό ενώπιον των ηγετών της Ευρώπης στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου που θα εστιάσει τα θέματα έρευνας και καινοτομίας. Πρέπει να βρούμε μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν υποστήριξη στο δυνατό υψηλότερο επίπεδο ώστε να γίνει ένας φάρος πρωτοπορίας η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα και την καινοτομία. Κομβικό και ζωτικό είναι αυτό το σχέδιο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ υποστηρίζω το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας δώσει μεγάλη υποστήριξη στην κατεύθυνση αυτή ώστε να είναι επιτυχές το σχέδιο αυτό. Η συγκεκριμένη μας στόχη είναι η εξή. Να εστιάσουμε την έρευνα και την καινοτομία στις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας μας που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη και ο κόσμος, που είναι και κύριες προτεραιότητες για τους λήπτες αποφάσεων και που συγχρόνως έχουν παρουσιάζουν ευκαιρίες αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, κλιματική αλλαγή, ασφάλεια ενέργειας, τροφιμική ασφάλεια, υγεία και γύρανση του πληθυσμού. Το να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε λοιπόν όλα αυτά τα εμπόδια για την πλήρη κυκλοφορία τη πληροφορία και τη δημιουργία μια ενιαίας αγορά για την έρευνα και την καινοτομία είναι ο στόχο μα. για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι καινοτόμε εταιρείε, ιδίω οι μικρομεσαίε εταιρείε έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση και ότι οι ελπιδοφόρε νέε ιδέε θα μπορέσουν να δοκιμήσουν στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Το σχέδιο μας θα βασίζεται σε μια ευρύτερη κατανόηση του τι είναι η καινοτομία. Φυσικά η καινοτομία βασίζεται στην έρευνα, αλλά που συμπεριλαμβάνει και άλλες μορφές, όπως παραδείγματος χάρη νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέους τρόπους διαχείρισης, νέα σχεδίαση και μάρκετινγκ και νέες υπηρεσίες. Θα καλύπτει κάθε στάδιο της αλυσίδας καινοτομίας από την αρχική σύλληψη εφιών ιδεών μέχρι την τελική του εμπορία για να λύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα που συνάπτονται με βασικές προκλήσεις της κοινωνίας. Το σχέδιο αυτό θα καθορίσει μια σειρά από στρατηγικούς στόχους που θα λέγονται οι ευρωπαϊκές σχέσει σχέσεις καινοτομίες, ώστε να φέρουμε κοντά τα προγράμματα μας έρευνα και ανάπτυξη μαζί με μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την ζήτηση, όπως είναι δημόσιες αγορές, τυποποίηση και ρύθμιση. Θα είναι φιλόδοξο λοιπόν τόσο για την εμβέλειά του όσο και για την έκτασή του το σχέδιο αυτό δεν θα είναι πρόσθετα σχέδια κοντά στα υπάρχοντα, όπως είναι οι κοινέ πρωτοβουλίες τεχνολογίες λοιπά, οι εταιρικέ σχέσεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, η, αγορά των, η πρωτοβουλία των αγορών και η τεχνολογία πληροφοριών. Αντίθετα, θα χρησιμοποιήσει αυτέ τι πλατφόρμε στο σχέδιό μα και θα τι ολοκληρώσει όπου δει. Υποστηρίζω λοιπόν όλα αυτά τα μέτρα για να μπορέσουμε να, να ευνοήσουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα έρευνα και επιστήμη καθώ και καινοτομία. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το κεφάλαιο κινδύνου, το Ευρωπαϊκό αυτό ταμείο, θα μπορούσαν να έχουν ένα σημαντικό ρόλο για να χρηματοδοτήσουν προγράμματα στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει το στόχο του 3% χρηματοδότηση σε επίπεδο ΑΕΠ για την έρευνα και την ανάπτυξη, που είναι ένα από του στόχου του προγράμματο Ευρώπη 2020. Είναι και ο κατάλληλο χρόνο επίση να προχωρήσουμε σε μια διαθεσμική συμφωνία και συζήτηση προηγουμένω για την απλοποίηση. έρευνα και η ανάπτυξη βρίσκονται στην καρδιά τη πρωτοβουλία Ευρώπη 2020. Η ναυαρχίδα κατά κάποιο τρόπο τη πρωτοβουλία μα θα πρέπει να είναι η επίτευξη διαφάνειας, σταθερότητος κανόνων, συνεκτικότητος, ταχύτητος και οκίτητος και επιτυχίας των διοικητικών διαδικασιών. Η καλύτερη χρηματοδότηση λοιπόν στον τομέα της καινοτομία σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε την εμπιστοσύνη και καλύτερο έλεγχο και να αποφύγουμε τους περιττούς κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δραστηριοποιήσει. Θέλουμε μία συμπεφωνημένη συμμετοχή όλων και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τη χρηματοδότηση της έρευνας. Ο κύριος στόχος της ανακοίνωσης απλοποίησης, η οποία θα εγκριθεί επίσημα αύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει μια διαθεσμική διαβούλευση για τα θέματα αυτά. Μέσα στην ανακοίνωση τα στοιχεία της απλοποίηση θα παρουσιαστούν σε τρει κύριες πλεξούδες. Η πρώτη από αυτές αφορά τα μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν βάσει του τρέχοντος νομικού πλαισίου. Το δεύτερο, η δεύτερη πλεξούδα θα αφορά τις αλλαγές στους κανόνες, αλλά με την διατήρηση της, του, των τωρινών συστημάτων σε ό,τι αφορά τις ζωές και το κόστος. Η τρίτη πλεξούδα αφορά τις δυνατότητε για μια εκβάθρον αλλαγή του υποδείγματος χρηματοδότησης, ώστε να προχωρήσουμε σε καταποκοπή χρηματοδότηση για συγκεκριμένα σχέδια. Η αναφορά στην ανάγκη πρόληψης απατών και στις στρατηγικές ανιχνεύσεων περιλαμβάνονται μέσα στην ανακοίνωσή μας. <clears throat> Η ανακοίνωση αυτή δεν αποτελεί νομοθετική πρόταση, αλλά μονάχα εναλλακτικέ λύσεις για την διαβούλευση και τη συζήτηση. Η συγκεκριμένη εκτίμηση κινδύνου και στρατηγικών θα είναι τμήμα της ε, τη αξιολόγηση αντικτύπου για μια μελλοντική νομοθετική πράξη. Όπως είπα και στην ακρόαση με ενώπιον του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο, εγώ θα υποστηρίξω πλήρως τι πρωτοβουλίε αυτές που έχουν σε στόχο να συνδέσουν τα εθνικά προγράμματα με αποτέλεσμα να υπάρξει καλύτερη συνεργασία των εθνικών προγραμμάτων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη, διότι θα πρέπει να συνενώσουμε του πόρου μα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει στην κοινωνία μα που κανένα κράτο μέλο δεν μπορεί από μόνο μεμονωμένο να αντιμετωπίσει. Μια περιοχή έρευνα για την Ευρώπη μπορεί να δημιουργηθεί και μονάχα αν υπάρχει πλήρη δέσμευση από όλα τα κράτη-μέλη. 95% όλη τη χρηματοδότηση στον τομέα τη έρευνα, καινοτομία και επιστήμη έρχεται κατευθείαν από τα 27 κράτη-μέλη. Αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε να υπάρξει περιττή επικάλυψη και κατακαιρματισμό των ερευνητικών προγραμμάτων και προσπαθειών για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τι ευκαιρίε που είναι διαθέσιμε για προγράμματα έρευνα τα οποία υποστηρίζουν από το δημόσιο τομέα στον τομέα τη έρευνα, τη επιστήμη και τη καινοτομία. Χαιρετίζω τι πρωτοβουλίε τη Ισπανική Προεδρία κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου για να προωθηθεί το θέμα της αύξησης κινητικότητας των ερευνητών και της ανάγκης βελτίωσης της κάλυψης σε κοινωνικό επίπεδο από κοινωνικές παροχές των ερευνητών. Για τους στόχους αυτούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στοχευμένες ε, στοχευμένα εργαλεία μέσα στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και αυτό επιτρέπει καλύτερη διαδικτύωση και συνεργασία μεταξύ εθνικών προγραμμάτων. Τα εργαλεία αυτά πηγαίνουν από το σχέδιο Ειρήνες, το οποίο βελτιώνει τις δυνατότητες διαδικτύωσης και φτάνω στα μέτρα του άρθρου 158 που αφορούν την πλήρη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινά προγράμματα μαζί με κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη. Πέρυσι τα κράτη-μέλη προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω και προχώρησαν σε μια πολιτική διαδικασία κοινού σχεδιασμού για την έρευνα αυτή η κοινή μορφή σχεδιασμού είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών μελών με την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν κύριε προκλήσει τη κοινωνία μέσα από κοινέ έρευνε, κοινέ ερευνητικέ δράσει που υποστηρίζονται από το δημόσιο τομέα. Πριν από λίγο, στι 15 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την πρώτη πρωτοβουλία προγραμματισμού για να αντιμετωπίσει μεγάλε προκλήσει, ξεκινώντα μια μεγάλη στρατηγική έρευνα σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίσει νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως Πάρκινσον, Alzheimer και κάποια άλλη που ξέχασα. Η Ευρώπη λοιπόν έχει να παίξει σημαντικό ρόλο μέσα στη στρατηγική του 2020. Έχει εγκρίνει τρεις νέες πρωτοβουλίες για κοινή σχεδίαση που περιλαμβάνουν την ε, τροφιμική ασφάλεια, την ασφάλεια στη γεωργία, κλιματική αλλαγή, πολιτιστικά κληροδοτήματα και επίσης την ανάγκη να έχουμε μια υγεία μια υγιή δίαιτα για υγιή ζωή. Όλα αυτά θα είναι η, θεμέλη, η δομική λύθη της πολιτικής μας, η εφαρμογή της Ένωσης για την Κοινοτομία θα μας επιτρέψει να έχουμε μια καλύτερη χρήση της κοινή σχεδίασης και να τη συναρμόσουμε με άλλα εργαλεία πολιτικής. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι το μεγαλύτερο δημόσια χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα στον κόσμο. Η απόφαση του 7ου προγράμματος πλαισίου προβλέπει για το 2010 να γίνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ανεξάρτητη και πλήρη αποτίμηση της εφαρμογής του 7ου προγράμματος πλαίσιου μέχρι στιγμής. Η ομάδα πυρογνωμόνων για αυτό το στόχο θα, θα εξετάσει την βάση τον τρόπο εφαρμογής και τα αποτελέσματα του 7ου προγράμματος πλαισίου και θα βασιστεί σε ένα ευρύ φάσμα στοιχείων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται στατιστικές λεπτομερείς για την εφαρμογή εξωτερικές μελέτες, ε, συνεντεύξεις και αναλύσεις και άλλες μελέτες. Θέλουμε να ανατάμουμε τις θετικές και αρνητικές πτυχές του προγράμματος αυτού, να δούμε πού είναι τα ισχυρά και τα ασθενή σημεία του, να δούμε ποια λειτουργούν καλά, ποια λειτουργούν λιγότερο καλά και να δούμε πού μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Επίση, θα εξετάσουμε πώ μπορούμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Όπω και τα μέλη τη Επιτροπή σα, εγώ ανησυχώ για το γεγονό ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν συμμετέχουν επαρκώ στα προγράμματα αυτά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει στο μέλλον. Η τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνώμων θα δημοσιευτεί το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αν θέλει ο Θεός. Η Κομισιόν τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο θα δώσει μια πλήρη απάντηση στα αποτελέσματα, στα πορίσματα των εμπειρογνώμων και αυτή η κομισιον το στη το δεκεμβριο θα συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν κλείσω την παρουσίασή μου, με μεγάλη χαρά θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι οι επιστήμονες από το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα είναι παρόντες 4 με 6 Μαΐου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα παρουσιάσουν μια έκθεση για τι ερευνητικέ προόδου σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων. Είμαι σίγουρη ότι τα μέλη τη Επιτροπή σα, κύριε Πρόεδρε, θα είναι σε θέση να είναι παρόντε στην έκθεση αυτή και να δούνε από πρώτο χέρι τι σημαντικά πράγματα κάνει το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για το τελευταίο που είπατε. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει πράγματι κάποιο από αυτή την πρωτοβουλία, ο οποίο έχει προσκληθεί να παρουσιάσει τα θέματα αυτά και θα συζητήσει μαζί μα. Αλλά τώρα θα ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση με την κυρία Επίτροπε. Ο κύριο Τζαβέλα. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο για την παρουσία της εδώ σήμερα. Είναι τιμή μας ε, και μας διαφωτίζει η παρουσίαση του προγράμματος για την έρευνα και την ανάπτυξη. Για την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία δεν υπάρχει μετρικό σύστημα προς το παρόν ε, για τις αποδόσεις και τις ε, ε, και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ε, κατά την εφαρμογή της Ευρωενωσιακής Πολιτικής για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Μετά τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αξιολόγηση του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει διαρκώς ότι χρειάζεται μια πιο συνεκτική και συστηματική χρήση των ε, δικτών που βασίζονται σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Επιπροσθέτως, έχει εκκινηθεί η πρωτοβουλία Start Metrics ε, για τη μέτρηση ε, των της επιστημονικής απόδοσης των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης με αυτά ως δεδομένα σύμφωνη το ότι πρέπει να υπάρχει ένας ε, μηχανισμός για την αξιολόγηση που θα βασίζεται σε ε, βάσεις δεδομένων ε, ώστε να βοηθηθούμε και να μπορέσουμε να καταρτήσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο υπάρχουν 8 και άλλες σχετικές πολιτικές. Επίσης μιλήσατε για τον κοινό προγραμματισμό. Δεν πιστεύετε ότι σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωσης και είπα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ε, προάγοντας έτσι έναν διατλαντικό χώρο έρευνας και ανάπτυξης. Ο κύριος Σοντή, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω ε, την Επίτροπο αναρωτιόσασταν αν θα καθόσασταν ε, στο Προεδρείο. Μα ε, κάνατε από τις καλύτερες ακροάσει σε σχέση με τους ε, υπόλοιπου επιτρόπους και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήταν άμεσά μας και πάλι. Για να αρχίσω θα έλεγα ότι διωγγώνονται διαρκώς τα προβλήματα με τους ελέγχους που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα ερευνητικά κέντρα. Η προσωπική μου άποψη όμως είναι ότι όλα βαίνουν αισίως. Ε, γιατί ε, σε κοινή ομάδα εργασίας με την ομάδα ελέγχου των προϋπολογισμών ε, παρακολουθήσαμε τις εργασίες των δύο επιτροπών και πιστεύω ότι αρχίζει να διαφαίνεται μια πολιτική συνένεση για να βρούμε μια διέξοδο το, η ανησυχία είναι να, να μην είναι πλέον δημοφιλής η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των κακών ελέγχων και κυρίως στους εθνικούς πολιτικούς κύκλους. Αυτό θα αποτελέσει πρόσκομο όταν κληθούμε να διαπραγματευτούμε με τα κράτη-μέλη για την ε, περαιτέρω, πώς να το πω, κοινοτικοποίηση των ε, ε, ερευνητικών κονδυλίων για τα επόμενα προγράμματα πλαίσιο. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι δεν μας ανησυχεί το μέλλον ε, γιατί θα ε, επιλέξουμε την απλούστευση αλλά πρέπει να κλείσουμε τους λογαριασμούς ε, του παρελθόντος τηρώντας τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Πρέπει να βρούμε μία διέξοδο. Μία ερώτηση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τι πιστεύετε για την προστασία ε, της επιστημονικής ε, έρευνας και για τη λειτουργία του ενιαίου Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Δεύτερη ερώτηση. Για την έρευνα στον ενεργειακό τομέα και κυρίως για τα, για τα στρατιωτικά προγράμματα, ε, θα θέλατε να σχολιάσετε αυτό το θέμα και τέλος. Είπατε ότι προεδρεύεται σε μια ομάδα εργασία επιτρόπων ε, για όλα τα ζητήματα που άπτονται της έρευνα. Ωραία. Η οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς, η βιομηχανική πολιτική και η πολιτική έρευνα πώς συνδέονται, με ποιο τρόπο μπορείτε να μας μιλήσετε ε, για την συνοχή που ε, πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις τρεις πολιτικές. Ο κύριος Γκέρεκ. Ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσεται συχνά υπέρ της ε, πολιτικής βούλησης ε, και παραμελεί τα απτά αποτελέσματα της έρευνας και της ανάπτυξης. Θα δώσω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για τα ε, θέματα των κλιματικών αλλαγών. Ε, δεχτήκαμε ένα σενάριο που είναι επικίνδυνο για την οικονομία μας. Καταπολεμούμε τις κλιματικές αλλαγές και θέλω να ρωτήσω δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικούς μας ε, επιστήμονες που θα μπορούσαν ε, στα πλαίσια ενός ε, κοινού προγράμματος να εξακριβήσουν αυτό το σενάριο σχετικά με την επίπτωση που έχει το διοξίδιο του άνθρακα επί των κλιματικών αλλαγών, αυτά που βλέπουμε δηλαδή στην τέταρτη έκθεση του IPCC. γνωρίζουμε ότι γίνονται επιστημονικές προσωμιώσεις, οπότε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την εξακρίβωση, κάτι άλλο τώρα. Ένα εξαιρετικά δαπανηρό πρόγραμμα, τον Καλλιλέο, ε, μπορεί τελικά να αναβαγίσει, έμαθα σήμερα, μα δεν έχουμε ε, ε, επιστήμονες, δεν έχουμε μηχανικούς εδώ. Για ποιο λόγο οι Ρώσοι ήδη έχουν το δικό τους GPS. Κάτι άλλο τώρα, προετοιμάζουμε διάφορα σχέδια συστάσεων και κανόνες για τις εκπομπές, για τις ανώτατες τιμές εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, φερρυπίν ναι, για τα οχήματα. Από τεχνικής πλευράς ε, είναι ανέφικτες οι συστάσεις μας, ε, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ακριβής ε, υπολογισμός μας λένε. Μήπως μπορούμε να βρούμε λοιπόν καλύτερες μεθόδους μέτρησης. Ε, κάτι άλλο τώρα. όλοι γνωρίζουμε πως πρέπει να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι τις βοηθάμε με τους κανόνες που έχουμε τώρα περί διανοητικής ιδιοκτησίας. Ευχαριστούμε ο Τσάρας τσίτσεστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, με τη σειρά μου να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Γκίγκαν Κίνε στην Επιτροπή μας. Ε, ζητώ συγγνώμη που αργοπόρησα και έφτασα στο μέσο της ε, παρουσίασής σας. Ε, ίσως ρωτήσω κάτι που ήδη αναφέρατε στην παρουσίασή σας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα μπορούσατε ίσως να αναπτύξετε περαιτέρω κάποια θέματα που ίσως έχετε αναφέρει. Όπως είπε ο κύριος Σοντή, προβλέπεται απλούστευση των κανόνων ε, και μπορεί ε, να αποτελέσει αυτό πρόσκομα για τις ε, μικρές οντότητες που θέλουν να συμμετάσχουν στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Μιλήσατε καθόλου για το πόσο μπορούμε να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, πρέπει να έχουμε αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο των ε, κονδυλίων ε, της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερο θέμα, η αριστεία. Αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, δηλαδή αν έχει σημειωθεί επιτυχία και αν με την αρχή της αριστείας έχουν βελτιωθεί τα ερευνητικά προγράμματα. Ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κυρίως το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συγγνώμη, έπρεπε να σας είχα δώσει ήδη το λόγο, αλλά δεν σας είδα. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να πάρουμε μέρος σε αυτό τον διαρθρωμένο διάλογο η έρευνα και ανάπτυξη είναι φυσικά τμήμα της καινοτομίας και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποια προβλήματα επικοινωνίας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και υπάρχουν ε, διάφορες προκλήσεις όπως η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, οι δημογραφικές αλλαγές, και το θέμα της συνεργασίας των δημόσιων επενδύσεων με τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα φτάνουν το 3%. Ε, αυτό είναι κάτι το εφικτό στις περισσότερες χώρες εκτός από τις λεγόμενες νέες χώρες. Ε, πέραν του 2% του ΑΕΠ δεν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε και αυτό γιατί δεν έχουμε ερευνητικέ δομές που θα μπορούσαν να προσελκύσουν επενδύσεις από ιδιωτικές επιχειρήσεις η έλλειψη υποδομών στον τομέα της έρευνας συνοδεύεται επίσης από τα προβλήματα που έχουν κληρονομήσει οι μεταβατικές περίοδοι μετά το κομμουνιστικό καθεστώς. Απαιτείται λοιπόν ένα πρόγραμμα δράσης για να αποκατασταθούν οι υποδαμές αυτές, έτσι ώστε να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τις επενδύσεις για τις οποίες ανήκει τις ευκαιρίες πλέον το, το πρόγραμμα, το 7ο, 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Να σας δώσω ένα σύντομο παράδειγμα το οποίο από μόνο του σας ε, δίνει να καταλάβετε ποιες είναι οι δυνατότητες των υποδομών. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Πολωνία έχουν διασφαλίσει περίπου 63 εκατομμύρια ευρώ από το 7ο πρόγραμμα από τον Οκτώβριο του 2008 για 50 προγράμματα. Ο πληθυσμός των χωρών αυτών ξεπερνά τα 67.200.000. Αν το συγκρίνει κανείς αυτό μπορεί να πάρει το παράδειγμα της Γαλλίας με πληθυσμό 63,8 εκατομμυρίων και με απορροφητική ικανότητα 570 εκατομμυρίων ευρώ για 365 προγράμματα κατά τη διάρκεια της ιδίας χρονικής περίοδου. Αυτό λοιπόν θέτει κάποια ερωτήματα. Πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα της έρευνας που θα πρέπει να αναδιορθωθεί σε ορισμένα κράτη-μέλη για να έχουν πραγματικά την ευκαιρία να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε ποσά του προγράμματος πλαισίου 7 και 8 θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο τα, τα, χρηματοδότηση των κρατών αυτών, δεδομένου ότι κινδυνεύουν να μην έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή έρευνα και πώς θα βοηθήσει η Κομισιόν τα κάτι μέλη να αναπτύξουν την ερευνητική του υποδομή. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Έχω τώρα πολύ κόσμο. Μήπως μπορούμε να είμαστε λίγο πιο σύντομοι στα ερωτήματά μας. Κύριε Κρυβάλιου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για το πάρα πολύ λεπτομεριακό πρόγραμμά σας που μας παρουσιάσατε. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια όμως. Ξέρω ότι ο στόχος σας είναι η καινοτομία και η πρόθεσή της, αλλά θέλω να λάβετε υπόψη και την κοινωνική καινοτομία. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια η οποία πρέπει να περιληφθεί στον ορισμό της καινοτομίας. Σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της χρηματοδότησης της έρευνας, εγώ αναγνωρίζω το γεγονός ότι έχετε διαχωρίσει ορισμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν καθ βάσει των τωρινών κανονισμών και αυτά που χρειάζονται μια ριζική αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό είναι μια καλή και αρκετά ρεαλιστική προσέγγιση, γιατί έτσι κάποια από αυτά τα μέτρα μπορούν να εγκριθούν και να εφαρμοστούν αμέσως. Αυτό μας συνδέει με το ζήτημα το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, το εργαλείο για τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο. Για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα χρειαζόμαστε μια μεγάλη αποποίηση στα εργαλεία τα οποία αναφέρατε. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκα αυτή τη στιγμή, έχουν χρησιμοποιηθεί αλλά με δυσκολίες. Και υπάρχει ένας μείζον ρόλος απλοποίησης από την πλευρά της Κομισιόν στα εργαλεία αυτά τα οποία υπόκειται σε κοινό προγραμματισμό. Η τελευταία μου παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μετατρέψει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε εμπορεύσιμη οικονομική αξία, αλλά δεν έχουμε καινοτομία χωρίς έρευνα και ανώτατη παιδεία που είναι θέματα περιθωριακά ίσως λιγάκι στο, στο χαρτοφυλάκιό σας. Χρειαζόμαστε αριστεία λοιπόν στην έρευνα και επομένως θα πρέπει η Κομισιόν να έχει πάντα στο μυαλό της ότι η έρευνα εχμής πρέπει να παραμείνει μια προτεραιότητα και δεν το είπατε αυτό το πράγμα. Δεν τονίσατε ότι το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο και συναφείς πρωτοβουλίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν την άποψή σας για αυτά για τις μελλοντικέ κατευθύνσεις. Ο κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ. Επίτροπε, θα επαναλάβω κάποια από αυτά που είπα χτες όταν ε, συναντήθηκα με διάφορους κατασκευαστές ε, την ε, μετα, εκπροσώπους μεταποιητικής βιομηχανίας. Συγγνώμη. Ε, θα πρέπει να έχουμε κοινωνικούς στόχους, αλλά είναι περιορισμένοι κρίνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιορισμένοι γιατί έχουμε λιγοστούς πόρους για την έρευνα και δεν μπορούμε να τους σκορπίσουμε σε πληθώρα πρωτοβουλειών και προγραμμάτων. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και θαραλέοι για να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Ε, επίσης, ε, δεν θέλουμε τη δεύτερη θέση. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατεχεί η ηγετική θέση. Οπότε τον πύχη πρέπει να το θέσουμε ψηλά ε, και όχι σε μέσα επίπεδα ή χαμηλά. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι θα πρέπει η βιομηχανία μας να βασίζεται στην έρευνα και Φυσικά έχουμε δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση κατά 20%. Ωραίο αυτό, δεν θα ανταλλάξουμε, αλλά θα πρέπει να υπερβούμε αυτό τον στόχο. Αν τα δεν τα καταφέρουμε, δεν τα καταφέραμε, αλλά τουλάχιστον να έχουμε υψηλούς στόχους, ε, δηλαδή να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Ενεργειακή αποδοτικότητα τώρα στη στρατηγική 2020. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και βασικές πρωτοβουλίε. και ό,τι έχει σχέση επίσης με τη γύρανση του πληθυσμού έχει και σημασία. Ε, θέλουμε να ε, βασιστούμε στις λύσεις ε, και όχι να ασχολούμαστε με τα επιμέρους τμήματα της πολιτικής. Ε, για την απλούστευση, για τη χρηματοδότηση δεν διαφωνούμε. Θα ήθελα να τονίσω τώρα κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανταμοιβή τη καινοτομία, ε, για το οποίο χρειάζεστε φυσικά τα δικαιώματα ε, διανοητική ιδιοκτησία, αλλά δεν θα πρέπει να τα ερμηνεύουμε με στενό τρόπο, διότι έτσι τα αποτελέσματα της έρευνας ε, μένουν κλειδωμένα στα συρτάρια και δεν χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της έρευνας. Χρειαζόμαστε ισορροπία λοιπόν και πρέπει να έχουμε ανοιχτό πνεύμα, να βρούμε την ισορροπία δηλαδή ανάμεσα στα αποτελέσματα και την προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, και επειδή είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί σας, ε, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω γιατί πιστεύω ότι και εσείς ακολουθείτε τη σωστή κατεύθυνση. Η Αγγελική Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ κυρία Επίτροπε για την παρουσία σας και έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την ε, ακροασή σας. Είχατε δείξει το πόσο είσαστε προσιλωμένοι στην πρόθεση των θεμάτων έρευνας τότε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα. Καταρχήν χαίρομαι ότι αύριο θα προωθήσετε ήδη την ανακοίνωση αυτή για την ε, απλοποίηση. Δεν ξέρω το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία από τη δική σας πλευρά και επίσης αυτό συνδέεται με το θέμα που έθεσε ο κύριος Τσίτσεστερ για την απογραφειοκρατικοποίηση και αυτό το οποίο τόνισε ο κύριος Σόντι ότι στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, ιδίως αυτές που αναφέρονται στους κανόνες χρηματοδότησης και ελπίζω ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει σε όλα τα διάφορα εργαλεία, πρωτοβουλίες και σχέδια της ε, έρευνας να υπάρξουν ενιαία μοντέλα διαδικασίας και διαχείρισης και όχι κάθε πρόγραμμα να υπόκειται σε νέους κανόνες. Δηλαδή εναρμόνιση στο βαθμό του δυνατού των διαδικασιών και επίσης στο βαθμό του δυνατού απλοποίησης. Όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ θετικά για την κοινότητα των ερευνητών στην Ευρώπη. Δύο ακόμα σημεία θέλω να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, ταξιδεύοντας έξω από την Ευρώπη, βλέπω πάντα ότι δεν υπάρχει μια τόσο, δεν τόσο ελκυστικός ο ευρωπαϊκός ερευνητικός χώρος όπως θα θέλαμε. θέλαμε να φέρουμε στην Ευρώπη τους καλύτερους εγκεφάλους του κόσμου. Βλέπουμε όμως ότι δεν υπάρχει μεγάλη επιτυχία προσέλκυσης στην Ευρώπη, στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρ' όλα αυτά η ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα είναι πρώτης τάξεως δεν έχουμε απλώ όμω την κατάλληλη ακτινοβολία. Θα έπρεπε να κάνουμε επομένω κάποια προσπάθεια όλοι για να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία προ τον έξω κόσμο, ώστε να φανεί πόσο σημαντική είναι η έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε θα είμαστε πιο επιτυχείς στην προσέλκυση ταλαντούχων ερευνητών οι οποίοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στα προγράμματά μας. Επίσης, ό,τι αφορά τους ερευνητές, έχουμε προγράμματα όπως το Marie Curie, για παροχή υποτροφιών και πιστεύω ότι αυτά τα προγράμματα ε, ανταλλαγών και υποτροφιών όπως το Marie Curie παρέχουν ένα θαυμάσιο έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πρόταση σε σχέση με αυτά και επίσης σε ό,τι αφορά την κοινή πρόγραμμα, τον κοινό προγραμματισμό νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ε, πρωτοβουλία μετά από αυτά που ξέρω από τους εθνικούς ε, βουλευτές ξέρω ότι έχουν κάπως ε, κριτική στάση έναντι αυτών των κοινών προγραμμάτων και ορισμένοι νομίζουν ότι αυτά είναι μια μορφή παρέμβαση στην Ευρώπη στα εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Ίσως λοιπόν με τις συνθήκες της Λισαβόνας στην εφαρμογή τους και τη μεγαλύτερη παρουσία των εθνικών κοινοβουλευτικών θα μπορέσουν να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Κύριος Κλάντε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και εγώ έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για σας. Όχι μόνο για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο και την προετοιμασία του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην χώρα μου <clears throat> είχα την ευκαιρία να συναντήσω εμπλεκόμενους στην έρευνα εκπροσώπους από πανεπιστήμια, από ερευνητικά ιδρύματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλοι τονίζουν ακριβώς αυτό το θέμα της ε, απλοποίησης. Είναι ένα παράπονό τους εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δεν λένε συλλήβδιν, απλοποίηση, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα του φορολογουμένου πιάνουν τόπο. Και έχουμε ορισμένους οι οποίοι λένε ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκα τα συστήματα αυτά, άλλοι όμως λένε ότι είναι εφικτό να αντεπεξέλθει κανείς με αυτά τα μοντέλα διαχείρισης. Είναι χρήσιμο λοιπόν να έχετε επαφή με όλους, αλλά αν σκεφτούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πιο μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και οι πιο καινοτόμες και οι οποίες έχουν τρία ή πέντε άτομα, θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο μεγάλο είναι το άχθος το οποίο για αυτούς σημαίνει το να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία για να πάρουν τη χρηματοδότηση. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό της ερευνητικής χρηματοδότησης το οποίο αφορά ειδικά τις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις και να τεθεί κατά μέρος για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή του. Επειδή λοιπόν είναι σημαντικός ο καινοτόμος τους ρόλος, θα πρέπει να τους λάβουμε υπόψη και ένα παράδειγμα πριν από λίγου μήνε. κάποιος από αυτούς που είδα, του είπαν ότι ήσασταν σε, ένα, σε μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και απορρίφθηκε, η, απορρίφθηκε το πρόγραμμά σας γιατί από τους, έξι, ε, από τους έξι αξιολογητές οι πέντε δεν ήσταν και ο έκτος μονάχα μόνος του το απέριψε. Αυτό δεν είναι πολύ θετικό. Κύριε Τόγια. Ε, e- και από πλευρά μου θα ήθελα να σας καλωσορίσω Λυπάμαι που επιστρέφω σε ένα θέμα το οποίο έχει ήδη συζητηθεί από πολλούς συναδέλφους, αλλά θα κατανοήσετε ότι η ίδια ύπαρξή μας αποδεικνύει ότι είναι κεντρικό το θέμα αυτό, είναι το θέμα δηλαδή της απλοποίησης των λογιστικών κανόνων. Εγώ είμαι βουλευτής εδώ και πέντε χρόνια. Θεωρώ ότι οι καλύτερες ιδέες μας και οι καλύτερες πρωτοβουλίες όταν ακολουθούν δρόμους περίπλοκους, χωρίς λόγο περίπλοκους, χάνουν θα έλεγα την αποτελεσματικότητά τους και δημιουργούν έλλειψη αξιοπιστίας ή βάρος της Ευρώπης. Όλοι είμαστε υπέρ της άφησης των πόρων για την έρευνα. Θα πρέπει να συνοδεύεται όμως η μάχη αυτή που δίνεται για περισσότερα χρήματα με μια σοβαρή προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης. Χθες όλο το πρωί διοργανώθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον hearing και πήραν μέρος αρκετοί συνάδελφοι εδώ από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών. Εξετάστηκαν προσεκτικά τα βασικά προβλήματα που εντοπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ακούστηκαν και διάφορες ε, υποθέσεις για να επιληθούν τα προβλήματα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι λογιστικές, η συζήτηση είναι ανοιχτή, αλλά θα πρέπει κάποιος να κάνει το πρώτο βήμα. Η Επιτροπή μέσα από την ανακοίνωσή της μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, γι' αυτό σας ζητάμε να είσαστε πιο αποφασιστικοί. Υπάρχει λοιπόν ένα υψηλότατο επίπεδο προσδοκιών σε σχέση με τις ικανότητες τις οποίες έχετε και δύο μικρές επιμέρους σκέψεις να μου επιτρέψετε. Πρώτον, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν. Αν σαν παράδειγμα το αίτημα ένταξης σε ένα πρόγραμμα είναι τόσο περίπλοκο που μειώνει ε, τον αριθμό αυτών που κάνουν την αίτηση όχι μόνο ανάμεσα στις μικρομεσαίες αλλά και ανάμεσα στα ερευνητικά κέντρα. Θα πρέπει να το αλλάξετε βέβαια το σύστημα αυτό, θα πρέπει να απλοποιήσετε την κατάσταση. Όταν υπάρχουν προβλήματα ορολογίας θα έλεγα, ας προσπαθήσετε να το λύσετε όταν υπάρχουν προβλήματα ταξινόμησης. Όταν τα πληροφορικά συστήματα ανάμεσα στις γενικές διευθύνσεις είναι διαφορετικά, εξομαλύνεται την κατάσταση και μετά περνάμε στις ρυθμίσεις για τις διαφορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα λογιστικά συστήματα και μεθόδους. Και γι' αυτό ακριβώς και εγώ λοιπόν όπως και η συνάδελφος Νίμπλα υποστηρίζω τα κοινά προγράμματα γιατί και χρήματα περισσότερα θα μας δώσουν και σίγουρα το θέμα της συγκέντρωσης των πόρων το οποίο υπογραμμίσατε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να, κάθουμε, να πείσουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν ενιαία προγράμματα, σαν παράδειγμα το Ατσχάιμερ, αλλά για να το πετύχουμε πρέπει εμείς οι ίδιοι να είμαστε πιστικοί. Κύριος Μεσάρος. Ευχαριστώ την Επίτροπο που ήρθε στην Επιτροπή μας για να μας μιλήσει για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τις τελευταίες εξελίξεις ε, και το τι μπορούμε να περιμένουμε από το πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, θα θέλαμε να ε, ενημερωνόμαστε τακτικά και Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να έχουμε μια σαφή εικόνα σχετικά με τις δαπάνες, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων. Αυτή η αξιολόγηση έχει ζωτική σημασία και για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, κυρίως αν θέλετε ε, νέα καινοτόμα στοιχεία μέσα σε αυτό. Μας μιλήσατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη. Θέλετε να τους προσφέρετε μεγαλύτερη στήριξη, να μειώσετε το γραφειοκρατικό άχθος. Ε, προσυπογράφουμε πλήρως ε, αυτή τη θέση και αυτό ε, επιδιώκω εδώ και μία δεκαετία εξάλλου. Για την στρατηγική 2020 καλούμαστε να επομιστούμε πολλές νέες ευθύνες. Το πρωί με τον ε, Επίτροπο Ταζάνη μιλούσαμε για την ε, βιομηχανική παραγωγή και την ε, σημασία, την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλήσαμε για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν έχει δρομολογηθεί κάτι ε, για την έρευνα, ε, κυρίως ε, ως προς το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ η κυρία Εκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο για την παρουσία της σήμερα και για την στενή συνεργασία που έχει με την Επιτροπή το εκτιμούμε ιδιαίτερος. Βλέπετε πόσες ερωτήσεις, πόσοι συνάδελφοι θέλουν να σας υποβάλουν ερωτήματα ε, πολλοί συνάδελφοι ενδιαφέρονται για το χαρτοφυλάκιό σας ε, και θα έχουμε αγαστή συνεργασία στο μέλλον, ελπίζω. Ε, το τρίγωνο της γνώσης πώς θα διατηρηθεί, δηλαδή η έρευνα, η καινοτομία και η γνώση ε, και θέλετε να μειώσετε το γραφειοκρατικό άχθος. Ε, δεν θέλω να τετραγωνίσετε αυτό το τρίγωνο, αλλά θα ήθελα να μας μιλήσετε για κάποια προγράμματα στον ε, βιομηχανικό κλάδο, δηλαδή τα προγράμματα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα εργαλεία, παραδείγματο χάρη για τις κρατικές προμήθειες, ώστε να επιδείξουμε νέες τεχνολογίες και να ξεκινήσουν, να αρχίσουν να λειτουργούν μέσα στην αγορά. Δεύτερον, ε, πώς να ενδιαφερθούν ε, για αυτά τα θέματα οι νέοι. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό κριτήριο για την στρατηγική 2020 και το δημογραφικό μας ε, ζήτημα. Δεν θα έχουμε αρκετούς ανθρώπους στον τομέα της έρευνας εάν δεν καταβάλουμε συνειδητές προσπάθειες τους προσεχείς μήνες και χρόνια. η κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Χαίρομαι που έρχεστε να μας παρουσιάσετε τις νέες σας κατευθύνσεις στην τρέχουσα περίοδο νομοθετικών εργασιών. Κάνετε ένα απολογισμό και λέτε ποιες είναι οι νέες κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν. Στην τελευταία θητεία μας έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για την μείωση της γραφειοκρατίας και υπήρξε το πρόγραμμα Eurostars για τις ε, εμπλεκόμενες στην έρευνα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ υπήρξαν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω αυτού του προγράμματος που μπορούν με ταχείες διαδικασίες να πάρουν τη χρηματοδότηση και να ξεκινήσουν τις εργασίες τους. Είναι μικρές εργασίες, μικρές εμβέλειες εργασίες, οι οποίες όμως πράγματι μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά προγράμματα καινοτομία. Δημιουργούν με τον τρόπο αυτό και νέε θέσει εργασία και καινοτόμα αποτελέσματα. Δεύτερον, χρειαζόμαστε καλύτερη διαδικτύωση σε διεθνέ επίπεδο. Θα μπορούσατε να φανταστείτε να υπάρχει και η δυνατότητα να έχουμε ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν νέα πανεπιστήμια στον Περσικό κόλπο, τα οποία ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε τέτοιε ανταλλαγέ. Στην Κίνα επίση έχουν δημιουργηθεί 50 ή δημιουργούνται 50 νέα πανεπιστήμια στου τομεί αυτού. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν φοιτητέ οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε στην Κίνα και να σπουδάσουν και να έρθουν τούμπαλιν Κινέζοι φοιτητέ στην Ευρώπη. Θα μπορούσατε λοιπόν να το έχετε αυτό υπόψη σα σαν μια δυνατότητα ανταλλαγών. Τέλος, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, νομίζω ότι ένα βασικό στοιχείο θα πρέπει να είναι η έρευνα στην Γεωργία, όπου προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ένα πακέτο 50 εκατομμύριων ευρώ για την έρευνα στην υγεία διατροφή των ζώων, για τα υγιή τρόφιμα, για να έχουμε καθαρό νερό στην γεωργία, καθαρά προϊόντα κτλ. Θα έχουμε, έχουμε αύξηση του πληθυσμού συνέχεια στον πλανήτη μα θα έχουμε σύντομα άλλο ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων, ενώ μειώνονται σημαντικά οι αρρώσιμε εκτάσει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν και εδώ μια έμφαση στα τρόφιμα, στη γεωργία, στην ανεώσιμη ενέργεια και επίσης ένας άλλο τομέας σημαντικός είναι η αποδοτικότητα της ενέργειας. Εδώ προβλέπεται πάλι ένα πακέτο 50 εκατομμυρίων ώστε να έχουμε φτηνότερη και πιο αποδοτική ενέργεια για τους καταναλωτές μας. Ευχαριστώ. κυρία Θέλετε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στην κυρία Επίτροπο καταρχήν ότι την ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολος είναι ο ρόλος της. Έρχεται σε στιγμές διαταραχών, κλειδονισμών. Γιατί τα θέματα της έρευνας είναι τόσο ευραία ώστε σε εποχές κρίσης όλοι προσπαθούν να βάλουν χέρι στο προπολογισμό της έρευνας. Ξέρουμε ότι μέσα στις δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι σημαντική η έρευνα και ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια κοινοτική πολιτική, μια ενωσιακή καλύτερα πολιτική για την έρευνα. Αλλά υπάρχει μια πλειάδα απειλών εναντίον της έρευνας. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για σας η Γενική Διεύθυνση Έρευνα έχει ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή δομή και έχει ένα πρόγραμμα συνεργασία που κινητοποιεί ανθρώπινου πόρου. Έχουμε από τη μια μεριά τα νέα προγράμματα αυτά, αλλά τα νέα αυτά προγράμματα δεν θα δημιουργήσουν την αυξανόμενη ε, ανταγωνιστικότητα παρά μόνο με προγράμματα όπως αυτό της, ε, το πρόγραμμα Marie Curie και πρέπει να σας πω ότι αν οι Beatles με δύο κιθάρες και ένα συσσωρευτή μπόρεσαν να κάνουν μια επανάσταση στη μουσική, δεν χρειάζεται εμεί να χρησιμοποιήσουμε τόσο αβαρύγδουπα όργανα για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί ο 21ος αιώνας βρίσκεται υπό την αιγίδα της σκέψης και της πληροφόρησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία για να εργαστούμε καλύτερα. Και όλα αυτά τα οποία λέμε σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο 8 η συνεργασία δεν υπάρχει στο φύλλο φιλοπορία που βλέπω αυτή τη στιγμή για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Γι' αυτό θα ήθελα να σας, σας ρωτήσω, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε εμείς να επιτύχουμε μια πρόοδο, όχι στη μουσική, αλλά στην επικοινωνία παραγωγή χάρη, που με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να προσελκύσει του νέου και να του κάνει πραγματικού εμπλεκόμενου σε όλα αυτά τα θέματα. Πώ θα κινητοποιήσουμε του ανθρώπινους πόρου, Χρειάζεται λοιπόν καινοτομία. Σκεφτείτε να έχετε μια πραγματική καινοτομία στα θέματα αυτά τη επικοινωνία που συνάπτονται με την έρευνα για να κινητοποιηθούν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να καταλάβουν πού πρέπει να πηγαίνει η σκέψη και η έρευνα. Äh, Ίσως θα πρέπει να δώσουμε στην κυρία Επίτροπο την ευκαιρία να απαντήσει στις πολλαπλές και αρκετά διαφορετικές ερωτήσεις που τις απευθύνθηκαν μέσα σε ένα εύθετο και λογικό χρονικό διάστημα. Thank you, Chairman. Um, Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> Να αναφερθώ στον τελευταίο μιλητή, την κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες. Πράγματι η καινοτομία χρειάζεται και στη γενική μας διεύθυνση και γι' αυτό προσπαθούμε εγώ και η ομάδα μου για να μπορέσουμε να καινοτομήσουμε και στη γενική διεύθυνσή μας. Θα ήθελα να αναφερθώ στον στόχο του 3%. Πολλοί το έθεσαν αυτό. Κάποιες χώρες έχουν ανησυχίες γύρω από τα θέματα αυτά. Άλλοι είπαν ναι στο 1%, άλλοι στο 2% και προσπαθούμε να συμφωνήσουμε στο 2% και γι' αυτό το εξετάζουμε προσεκτικά για να μπορέσουμε να δώσουμε τους λόγους που θα εξηγούν την κατάσταση που ισχύει διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να πούμε ότι στο στόχο του 3% συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη τα οποία θέτουν τους δικούς τους στόχους. Αυτό το 3% δεν είναι θα έλεγα ένα παπούτσι που έχει ένα νούμερο και ταιριάζει σε όλους θα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των χωρών που δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο αυτό. Να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε συγκεκριμένους στόχους. Οι υπηρεσίες μου είναι σε στενές επαφές με όλες αυτές τις εθνικές διοικήσεις τις τελευταίες εβδομάδες για να τους βοηθήσουμε να ορίσουν ποιοι εθνικοί στόχοι θα είναι οι καταλληλότεροι να επιδιωχτούν χαρακτηρίζοντας με συγκεκριμένο τρόπο τις ανάγκες τους. Έτσι θα μπορέσουμε ουσιαστικά να κινητοποιήσουμε την επιδίωξη των εθνικών στόχων που να λαμβάνει υπόψη τα εθνικά επιμέρους χαρακτηριστικά. Για τους δείκτες. <clears throat> Έχω δημιουργήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που συνεργάζεται με την Γενική Διεύθυνση Έρευνας και με τη Γενική Διεύθυνση για την οποία είναι υπεύθυνο ο Επίτροπος Ταγιάννη και τον προϋπολογισμό επίσης. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε συστήματα δικτών για το τι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτά τα συστήματα δικτών. Για να το εξετάσει κανείς αυτό με ανεξάρτητο τρόπο και εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή δημιούργησε αυτές τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων αποτελούνται από καινοτόμους επιχειρηματίες, είναι μια μικρή ομάδα, δεν είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου των κρατών μελών, αλλά νομίζω <clears throat> ότι θα οδηγήσουν σε νέες προτάσεις για την καινοτομία, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις ανάγκες καλύτερα. Γνωρίζουμε ποιο είναι το input, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα που βγαίνει από αυτό. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ήταν απογοητευτική. Πρέπει να λύσουμε επιμέρους προβλήματα όπως οι υποδομές για τις επενδύσεις, τα IPR γενικά ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τη βιομηχανία στην οποία εμπλέκονται. Οι γεωργοί έχουν μια συγκεκριμένη άποψη, αν ασχοληθείτε με το ICT έχουν επίσης διαφορετική άποψη. Όλες αυτές λοιπόν οι απόψεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτό είναι κάτι ε, στο οποίο θα ενδιαφερθεί πολύ, για το οποίο θα ενδιαφερθεί πολύ αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά αποκλειστικά τον δικό μου τομέα, αφορά σαφώς και τον τομέα του Μπαρνιέ, του Επιτρόπου Μπαρνιέ και θα ήθελα να πω επίσης ότι αυτό το στόχο έχει η ομάδα της Επιτροπής που δημιουργήθηκε. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι χρειάζεται να γίνει έτσι ώστε όταν έχουμε τα στοιχεία προς δημοσίευση, τα στοιχεία αυτά να είναι φιλόδοξα, να θέτουν στόχους πιο σημαντικούς από ό,τι στο παρελθόν και ο κόσμος να συγκινηθεί σε εισαγωγικά, να πούνε ότι να λοιπόν έχουμε υλικό για να προχωρήσουμε. Και κάθε τμήμα του προγράμματος αυτού, το οποίο θα ανήκει σε διαφορετικούς επιτρόπους, θα προωθηθεί με τον σωστό τρόπο. Τα πράγματα δεν είναι συνηθισμένα θα έλεγα. Όλοι οι επίτροποι τα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτό και εγκάρσια έτσι ώστε να μην αφήσουμε τίποτα απ' έξω. Το θέμα των δημοσίων προμηθειών είναι επίσης σημαντικό θέμα και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Οι υποδομές για τον τομέα της έρευνας. Άκουσα αυτά τα οποία είπατε για τις υποδομές της έρευνας στις νέες χώρες μέλη. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς βουλευτές γύρω από το θέμα αυτό. Ο κύριος Χάν, ο Επίτροπος Χάν, που ήταν και αυτός ερευνητής, γνωρίζει ποιες είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν. Έχει αρκετά χρήματα στη διάθεσή του, 85 δις συνολικά. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά με σωστό τρόπο πράγματι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η επιστημονική αξιολόγηση των, των προγραμμάτων τα οποία κατατίθενται προς αξιολόγηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και η αντικειμενικότητά μας επίσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να τα βελτιώνουμε. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει θα προσπαθήσουμε οι μικρομεσαίες να λειτουργήσουν σε ένα πολύ πιο ευνοημένο περιβάλλον, ευνοϊκό συγγνώμη περιβάλλον, είτε είναι μικρές επιχειρήσεις, ελάχιστες επιχειρήσεις, είτε είναι επιχειρήσεις διεθνικές, πολύ μεγαλύτερες, όλες αντιμετωπίζουν προβλήματα και πάντα παραπονούνται για την έλλειψη χρηματοδότησης. Είχα μια καλή συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων την προηγούμενη εβδομάδα. Έθεσα το θέμα στην τράπεζα. Μέσω του EIF έκαναν πράγματα τα οποία απεδείχθησαν θα έλεγα πολύ χρήσιμα. Η πρωτοβουλία θα έλεγα αυτή η κατανομή του κινδύνου είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί βλέπουμε ότι ομάδες εταιριών συνεργάζονται και από κοινού αναπτύσσουν μεγάλα προγράμματα υποδομών. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν πώς εμείς θα μπορέσουμε είτε να βρούμε ένα άλλο μέσο είτε να μετατρέψουμε το μέσο αυτό για να καλύψουμε τις ανάγκες μας για την απλοποίηση. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε ο κύριο Σόντι για τη μεικτή ομάδα εργασία ανάμεσα στην Επιτροπή σα και την Επιτροπή Ελέγχου προπολογισμών. <clears throat> Ήμουν στο ελεγκτικό συνέδριο για 10 χρόνια και γι' αυτό παρακολουθούσα τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών. Και υπάρχουν ε, πάρα πολλές μορφές δισταγμού γύρω από τις πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνονται για να αλλάξουν τα πράγματα. Όλοι θα πρέπει να έχουμε σαφείς οικονομικές βάσεις για να κρίνουμε και τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου να χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό, ουσιαστικό και σωστό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν με πάρα πολύ ενδιαφέρον περιμένω τις εξελίξεις των εργασιών σας. Στην ανακοίνωση και στη συνεργασία των επιτρόπων που ασχολούνται με την έρευνα προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τους κανόνες που έχουμε στη διάθεσή μας για να ερμηνεύουμε σωστά ε, τους κανόνες, να έχουμε σωστή ε, ελεγκτική διαδικασία και ε, εύκολες και μεμονωμένες δυνατότητες αίτησης συμμετοχής. Πάντα για την απλοποίηση. Τα μέσα θα επανεξεταστούν όταν έχουμε προχωρήσει στην διάμεση ε, αξιολόγηση να δούμε τι έχει πάει καλά και τι όχι. Και ελπίζω ότι έχουμε, θα έχουμε μετά το καλοκαίρι, μετά τους καλοκαιρινούς μήνες κάποιες πρώτες εντυπώσεις για τα προφίλ των ερευνητών. Εμείς θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να έχουμε συγκεκριμένους ρόλους, πρότυπα. Και εννοώ με αυτό. Κάθε φορά εκεί που πάω ο κόσμος μου λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας τους ε, μηχανικούς που θέλουμε, τους επιστήμονες που θέλουμε, δεν μπορούμε να τους βρούμε. Μπορείτε να μας βοηθήσετε, μπορείτε να μιλήσετε με τα κράτη-μέλη και τις αρχές για να έρθουν σε επαφή με τα πανεπιστήμια και να βρούμε, εν πάση περιπτώσει, συγκεκριμένα ρόλους με τους οποίους να ταυτιστούν οι νέοι επιστήμονες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επισκευάζουμε σε εισαγωγικά τη στρατηγική που ακολουθούμε προς την κατεύθυνση. Ελπίζω να συνεργαστούμε με την ερευνητική κοινότητα για να υπογραμμίσουμε τα μοντέλα, τα πρότυπα αυτών των ανθρώπων που από μικρή ηλικία έφτασαν μέχρι και να κερδίσουν τεράστια βραβεία επιστημονικά. including in the actual list that I Εγώ δεν σας έδωσα πολλές λεπτομέρειες και καταλόγους σε αυτά τα οποία είπα προηγουμένως λόγω έλλειψης χρόνου. Η κοινωνική καινοτομία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας και όταν μιλάμε για κοινωνική καινοτομία δεν μιλάμε μόνο για μία ή δύο πλευρές, μιλάμε για συνολικές παρεμβάσεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πόσο θα προχωρήσουμε στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας να δούμε πώς τα μέλη της Επιτροπής σας κύριε Πρόεδρε μπορούν με συγκεκριμένο τρόπο να δώσουν συμβουλές στον τομέα αυτό ή και σε άλλους τομείς. Γιατί εμείς ε, επιμένουμε στον ρόλο της κοινωνικής ε, καινοτομίας, όπως επίσης και ο πρόεδρος Μπαρόσο και η συμβουλή του. Ένας νέος τομέας και απαιτούνται νέες έρευνες. Θα πρέπει οι ερευνητές να βγουν από τα γραφεία και να επιστρέψουν στα εργαστήρια. Απαιτείται να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στους εμπλεκομένους στις διαδικασίες και μια σωστή κατανομή των κινδύνων. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να δει κανείς ποιες θα είναι και οι αναθεωρήσεις οι οποίες θα υπάρξουν στο τέλος του μήνα Μαΐου. Ο αρμόδιος επίτροπος έχει παραδεχθεί τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την πνευματική ιδιοκτησία, για την ευαισθητεχνία μάλλον. Πιστεύουμε ότι απαιτείται να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ευαισθητεχνία τώρα και ο κύριος Μπαρνιέ προσπαθεί να συνεχίσει την προσπάθειά του προς την κατεύθυνση αυτή. Απαιτείται όμως να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι ένας από τους επιτρόπους που συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα και θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. πολιτική στον επιστημονικό τομέα, αναφέρθηκα σε αυτό στην εισαγωγή μου, προγράμματα επίδειξης, και επιμονή στο πρόγραμμα 2011 στη μεταφορά τεχνολογίας, μεγαλύτερη πρόσβαση στις μικρομεσαίες και προγράμματα επίδειξης παράλληλα με το πρόγραμμα Blue Skies και άλλα. Ο κύριος Ρούμπικ είχε πει κάτι στο οποίο έχω ήδη απαντήσει. Συνεργάζομαι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δούμε σε ποιους τομείς μπορεί να μας βοηθήσει. Εγώ εμπλέκομαι στο πρόγραμμα ITER και στο μεγάλο θέμα της χρηματοδότησης του ITER. Θα σας κρατήσω ενήμερους για τις εξελίξεις. Θα ήθελα να πω όμως ότι εξ αρχής, στα πλαίσια της ανάγνωσης του φακέλου που είχα μπροστά μου, όλη η προσπάθεια την οποία έκανα είναι να θέσω το ITER σε ένα οικονομικό, θα έλεγα, υποστηρίξιμο πλαίσιο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σφαιρικό πρόγραμμα το οποίο ηγείται απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη σύνδεξη και τις δυνατότητες που παρέχει για την παραγωγή ε, ενέργειας καθαρής στο μέλλον, για την αντιμετώπιση ε, των αρνητικών συνεπειών της υπερθέρμανσης και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι σημαντικά για όλους. Οι ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν την προσοχή τους, τρέφουν την προσοχή τους στο ίτερ. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τους νέους υπολογισμούς κόστους για τη λειτουργία του προγράμματος, το οποίο θα πρέπει, όπως είπα, να είναι υποστηρίξιμο οικονομικά. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση σχετικά με το ίτερ αρχές Μαΐου, στις αρχές Μαΐου αυτή θα περάσει και από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και να είστε σίγουροι ότι προσπαθούμε και εγώ και οι υπηρεσίε μου συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες αρχές του προϋπολογισμού να βρούμε λύσεις οι οποίες να μην είναι βραχυπρόθεσμες λύσεις αλλά μακροπρόθεσμες που να βοηθήσουν την κατάσταση. Θα πρέπει να το δούμε αυτό και μαζί σας και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ίσως μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, για τα στοιχεία που μας δώσατε, τις πληροφορίες και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία μαζί σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελείωσε η συνεδρίασή μας. Σας παρακαλώ να αφήσετε την αίθουσα ταχαίως και γαληνίως γιατί θα ακολουθήσει μια συνεδρία των συντονιστών. Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσουμε.